Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Please. Καλημέρα συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Καθίστε για να ξεκινήσουμε. What is this song? The first item on the agenda is, as always, the adoption of the draft agenda. Can it be adopted? Fine. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνείτε, ωραία. Και μετά έχω να σας ανακοινώσω κάτι ε, λυπηρό. Ε, αυτό είναι το γεγονός ότι η Κλέρ Γκέντα που εργάστηκε μαζί μας εδώ και αρκετά χρόνια και ε, πριν έρθει στη γραμματεία ήταν στο τμήμα πολιτικής και σε άλλες επιτροπές, θα φύγει από τη γραμματεία το Μάρτιο. Η Κλέαρ ήταν μια εξαιρετική υπάλληλο, ε, πολύ καλός άνθρωπος, πάντα ε, προσέφερε στήριξη σε όλους, ε, υπεύθυνη για πάρα πολλά σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα τον όλο τομέα της πρόνοια των παιδιών και πραγματικά ε, λυπούμαστε πολύ που φεύγει και τη ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ε, επειδή είσαι ένα λαμπρό αστέρι βέβαια όλα θα πάνε πολύ καλά. <laughs> that was not for you this time. You need to do this by yourself, Αυτό δεν ήταν για σας, ήταν ε, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε διμερώς με την Κλέρ. Τώρα, στα διάφορα δεν έχω κάτι να σας πω. Και τώρα, σας παρακαλώ, προσδεθείτε, διότι Έχω πάρα πολλές ανακοινώσει να σας κάνω για τις αποφάσεις των συντονιστών ε, από τις συνεδρίε 23 Ιανουαρίου και θα αργήσουμε. Πρώτα-πρώτα, οι συντονιστές έλαβαν αρκετές αποφάσεις και θα πρέπει ε, για τα πρακτικά να τις αναφέρω όλες μία προς μία. Λοιπόν, αλλά έτσι έχει ο κανονισμός. Είναι το άρθρο 205. Λοιπόν, ε, αμφισβητούμενες συστάσεις εγκρίθηκαν ε, όπως προτείνεται από την Προεδρία για τις ε, διάφορες αναφορές. Ε, όλες είναι του 2017, θα σας λέω τον αριθμό. Είναι η 656, 657, 671, 702, 0712, 0715, 0727, 0728, 0792, 0808, 0835, 0943, 0956. Όλες θεωρήθηκαν παραδεκτές και έκλεισαν εκτός από τις 0792, 0943 και 0956 που θεωρήθηκαν μη παραδεκτές. Η αναφορά 0662 ε, επίσης το 2017 θα παραμείνει ανοιχτή και θα εξεταστεί μαζί με άλλες αναφορές ε, ε, για το ίδιο θέμα επιπλέον της σύστασης που έκανα και πάλι εγώ και για την αναφορά 0701 επίσης το 2017 αποφασίστηκε να ζητηθεί ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη διαβάσουμε στην Επιτροπή έμπλη ε, για γνωμοδότηση. Για την αναφορά 0705 αποφασίστηκε να ζητήσουμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την παραπέμψουμε και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για γνωμοδότηση. Η αναφορά 0720 αποφασίστηκε να διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Φάμα ΑΦΕΤ και ΝΤΡΟΑ για γνωμοδότηση και να τη στείλουμε και στην ΥΠΑΤΗ πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ε, πολιτική ασφαλείας. Η αναφορά 0775 αποφασίστηκε να ε, θεωρηθεί παραδεκτή, να εξηγήσουμε στον ε, αναφέροντα το περιεχόμενο του άρθρου 165 παράγραφος 1 και να προτείνουμε να στείλει καταγγελία στον ε, ε, Λετωνό συνήγορο του πολίτη και να θέσει το θέμα και στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λετωνίας και μετά να κλείσει. Για την αναφορά 0837 θεωρήθηκε παραδεκτή και αποφασίστηκε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω πληροφορίες και να στείλουμε την ε, αναφορά στην ΕΜΒΗ για πληροφόρηση. Τώρα, για την Καταλωνία, Έχουμε 29 σχετικές αναφορές, οι οποίες θεωρήθηκαν μη παραδεκτές βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφασίστηκε λοιπόν να ενημερώσουμε τους αναφέροντες για το άρθρο αυτό, το περιεχόμενό του και τη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου και να του στείλουμε ένα σύνδεσμο με τη συζήτηση για το θέμα της Καταλωνίας. Όλες οι άλλες αμφισβητούμενες συστάσεις εγκρίθηκαν όπως είχα προτείνει. Η κυρία Όκεν. Το ξέρω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλώς να γραφτεί για τα πρακτικά. Ότι οι πράσινοι, ε, υποθέτω και, για άλλους, δεν είχαμε την ευκαιρία ε, να το συζητήσουμε. Δεν είχαμε τίποτα γραπτό και χρειάστηκε να στείλω κάποιον άλλο στη συνεδρίαση και τελώ εν αγνία. Το ξέρω ότι πρέπει να λόγοδετούμε, αλλά αν είχα κάτι γραπτό πριν αποφασιστεί, θα μπορούσα ως συντονίστρια να κανονίσω την πορεία μου και να στείλω κάποιον, το Χωσέ Μαρία, κάποιον για να διαμαρτυρηθεί ή να εκφραστεί. λέτε ότι ήταν στο χρονοδιάγραμμα, αλλά και εσείς η ίδια ε, κάνετε αναδιατάξεις, αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα κτλ. Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα, απλώ να διαμαρτυρηθώ εντόνω και να γραφτεί στα πρακτικά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα το προσθέσουμε στα πρακτικά. Ε, να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία για τη διερευνητική αποστολή στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Okay, yeah, yeah, you may vote by raising. Ωραία, διαρατάσσω ε, στη χειρός. 20 με 22 ενάτου. Εγώ που έχω όμως την κάρτα ψηφοφορίας, όπως και οι υπόλοιποι, α χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματα. Already did it. I was a bit late on that. Μισό λεπτό. Έχω καθυστερήσει. That's it. So Marlene is raising her hand. Σηκώνει το χέρι της Marlene. Λοιπόν, εγώ έχω την κάρτα μου. Σύσταση 3α, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σύσταση 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σύσταση 4α, η τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σύσταση 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η σύσταση 5α, ε, η τροπολογία 5 δηλαδή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 7 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και 8 υπέρ, Against. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά σας παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is... Wait. The vote is now... After Mr. Mandel has voted it, I will... Αφού ψηφίσει και ο κύριος Μάντελ, τότε θα τελειώσει η ψηφοφορία. Okay, the machine seems not to be working. Δεν φαίνεται να δουλεύει το μηχάνημα. The card is not working. You can raise your hand and Καλά, σηκώστε το χέρι σας και θα τελειώσει η υπόθεση. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. The result is... Αποτέλεσμα. 20 υπέρ και μία ψήφος κατά. Λοιπόν, προχωρούμε στο σημείο 6 η ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε όσο γίνεται πιο διακριτικά. <laughs> Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Και παρακαλώ τους συναδέλφους να κάνετε όσο γίνεται περισσότερη ησυχία. Ε, μια εξερευνητική επιτροπή στη Λουσατία Λάουζιτ στη Γερμανία 14 με 16 Φεβρουαρίου ενεστώτος έτους. Και θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Τσάκη, με χαρά επικεφαλής τη αντιπροσωπεία Ευχαριστώ, Σεσίλια, για το λόγο. Επειδή έχουμε και διερμηνία, να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, την Ουγγρική. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας για την επίσκεψη αυτή και την υποστήριξη για το κείμενο που υπερψηφίσαμε μόλις για την Κύπρο. Νομίζω ότι ε, βοηθάμε τους Κυπρίους με την απόφαση μας αυτή. Έρχομαι τώρα στην αποστολή στη Γερμανία. Είναι πιο περίπλοκο το θέμα και πιο σύνθετο από αυτό που συζητούσαμε για την Κύπρο. Δύο είναι τα προβλήματα. Είναι πολύ ωραία αυτή η ε, περιοχή ανάμεσα στο Βερολίνο και τη Δρέσδη. Ε, είναι πολύ ωραίο μέρος και το τοπίο καταπληκτικό και είναι μια ωραία περιοχή για να μένει κανείς. Κατοικούν και πολλοί. Τι λέγουν λοιπόν οι κάτοικοι εκεί. Ότι είναι θεόσταλτο δώρο αυτό, αλλά ο διάβολος έχει βάλει στο υπέδαφος εκεί λιγνίτη έτσι κατά τη δημιουργία της πλάσης και του σύμπαντος. Και έχουμε ανοιχτά λιγνητορυχεία εκεί τα οποία ε, ε, ρηπαίνουν το περιβάλλον και πληγώνουν το τοπίο και αφήνουν και ουλές. Επίσης υπάρχουν 50.000 κάτοικοι εκεί που ανήκουν στη σοραβική εθνική μειονότητα. Δεν έχουν κράτος, έχουν δύο διαλέκτους ε, στην κοινότητά τους, εκεί των σοραβών και ορισμένες από τις ε, ε, εθνοτικές ομάδες έχουν υποστεί και εθνοκάθαρση ε, στο παρελθόν λόγω της εξορρεκτικής δραστηριότητας. Δηλαδή τους έχουν διώξει από εκεί και τους έχουν μεταφέρει σε αστικές περιοχές. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και παίζεται πολύ και η σορβική του ταυτότητα και ο πολιτισμός τους. τα μέλη λοιπόν αυτής της εθνικής μειονότητας αντιδρούν. έχουν υψώσει στη φωνή τους και έχουν ε, καταθέσει και μια τρίτη αναφορά για την προστασία της σοροβικής γλώσσας. Είναι δύσκολο το κείμενο να είναι ισόρροπο. Υπάρχει πρόβλημα γιατί δίστανται απόψεις. Ε, ο λιγνίτης που παράγεται εκεί χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτει το 1 τρίτο των αναγκών των ενεργειακών ε, Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει η δραστηριότητα από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι τέσσερα τα μεγάλα ε, εργοστάσια, μονάδες θερμοηλεκτρικές ηλεκτρικής παραγωγής. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι υπερσύγχρονα αυτά τα εργοστάσια. Αλλά ακόμα και τα υπερσύγχρονα δεν ε, αρκούν για να φιλτράρουν τελείως ε, τα αρούμενα ε, σωματίδια και να μην διαχέονται αυτά στην ατμόσφαιρα. Είναι τριπλάσια στατιστικά τα αναπνευστικά ε, νοσήματα και σε σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία ε, έχουμε και ρήπανση των επιφανειακών υδάτων και το pH ε, αποκλίνει από το φυσιολογικό pH του νερού. Λοιπόν, ε, είναι δύσκολη η κατάσταση. Τι θα κάνουμε εμείς, ποια είναι η σύσταση. Ε, που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε. Το γερμανικό κράτος να απαλύνει κάπως να ανακουφίσει τις συνέπειες της λιγνητικής δραστηριότητα εκεί και να ε, αφενός και αφετέρου να υποστηρίξει περισσότερο τους οραβούς, τη μειονότητα, την κουλτούρα τους και τον πολιτισμό τους. Για να είμαστε ειλικρινείς, η Γερμανία κάνει ήδη προσπάθειες και έχει σημαντικά ε, προγράμματα για την προστασία των ε, Υπάρχουν παντού δίγλωσες επιγραφές ε, στην περιοχή και πινακίδες ας πούμε. Δεν είναι τέλεια μεν η κατάσταση, αλλά ε, το αντιμετωπίζει η Γερμανία. Ο κόσμος ανησυχεί γιατί προβλέπεται να ανοίξουν άλλα δύο λιγνητορυχεία Και η ίδια η εθνική μειονότητα δεν συμφωνεί. Δηλαδή, αν γινόταν εκεί δημοψήφισμα, ο κόσμος θα ήταν διχασμένος, γιατί πρόκειται και για πολλές θέσεις εργασία. 8.600 είναι εργαζόμενοι στη λιγνητορυχία εκεί. Είναι καλοπληρωμένες θέσεις και η τοπική κυβέρνηση υποστηρίζει τα νοσοκομεία, τα σχολεία, γίνεται Μάλιστα και τα εργοστάσια και τα λιγνητορχεία υποστηρίζουν ε, την κοινότητα και οικονομικά. Πάντω κάποια στιγμή θα πρέπει να εγκαταλειφθεί αυτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω μία έκκληση αυτή τη στιγμή. Αν συμφωνείτε και αν συμφωνεί και η Πρόεδρος και οι συνάδελφοι, να στείλουμε μία επιστολή με ερωτήματα στη μόνιμη γερμανική αντιπροσωπεία και στη γερμανική κυβέρνηση δια του πρέσβη για να ρωτήσουμε ποια είναι η θέση της νέας ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε σχέση με τα λίγνη, και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Γιατί στο Πότσταμ έχουμε μέλη της ε, περιφερειακής κυβέρνησης εκεί της τοπικής του κρατηδίου ε, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης συναντήσει, εκπροσώπους της κοινότητας της ίδιας των Σοραβών αλλά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν την είδαμε. Προφανώς είναι τώρα μεταβατική περίοδος είναι υπηρεσιακή η κυβέρνηση και σχηματίζεται νέα, αλλά θα πρέπει να τη βολιδοσκοπήσουμε σε σχέση με τις προθέσεις της για τη συγκεκριμένη εξορρυκτική δραστηριότητα και βιομηχανία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την απάντησή τους, να οριστικοποιήσουμε το έγγραφό μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία και την ε, γραμματεία. Ήταν εξαιρετικές οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσει και η προετοιμασία όλη τη αποστολή εκεί. Ευχαριστούμε πολύ τη Γραμματεία. Ήταν πάρα πολύ καλή η διερευνητική αυτή αποστολή με καλά αποτελέσματα. Αλλά όπως σας είπα είναι τεράστια η περιπλοκότητα της κατάστασης. Εμείς προσπαθήσαμε να συλλέξουμε όσο γίνεται περισσότερες προφορίες για να είναι οι συστάσεις μας πολύ ισορροπημένες. Στο τέλος ευχαριστώ. Αυτά για σήμερα. Thank you very much. Very... Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον όπως πάντα και πολύ ακριβής η περιγραφή. Μάργαρετ Άουκεν, ευχαριστώ και σε ευχαριστώ και ένα Παλ. Ε, εξαιρετική πάντα η ηγεσία σου στις αντιπροσωπείες και το λέω και προς την ε, γραμματεία ε, και ε, προσυπογράφω όλα όσα είπες για τη γραμματεία. Μερικά πράγματα μόνο, πρώτο και κύριο, που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Υπάρχει σεβασμός εκεί ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Natura 2000, ε, οδηγία αντίστοιχη, ε, η οδηγία για τα ύδατα, για τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό δεν ήταν σαφές. Για θέματα περιβαλλοντικά δεν έχουμε πάντα πληροφόρηση και πολλοί αναφέροντες λένε ότι και οι ίδιοι δεν ενημερώνονται γιατί τα κρατάνε μυστικά τα στοιχεία. Αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων και κάτι που με ανησύχησε πάρα πολύ. Συγγνώμη Μάργαρετ αλλά κάτι τρέχει στην αγγλική καμπίνα. Να τα πω δανέζικα, λέει. Γιατί δεν αγγλικά μιλάω. Δεν ξέρω. Τι γίνεται με τη δανική καμπίνα σήμερα το πρωί. So, let's, let's see what happened to the English. Τι συμβεί τώρα με την αγγλική καμπίνα για να... Αφού αγγλικά μιλάω. Θέλετε να τα πω δανέζικα, τα πω δανέζικα. Μήπως σας βγουν καλύτερα. Nobody understands. So. Except you. Δεν, δεν καταλαβαίνει κανείς δανέζικα, εκτό από σένα, λέει η κυρία Άουκεν. Can I, can I ask the interpreters to make sure... Παρακαλώ τους διερμηνείς να φροντίσουν ότι είναι εντάξει οι καμπίνες και τα κανάλια τους. Μα αγγλικά μιλάει η ομιλήτρια. No, I'll take it in English here because I think that would be the easiest at least. Λοιπόν, εντάξει, συνεχίζω. Το Ξέρω ότι τα αγγλικά μου δεν είναι και τόσο καλά. Να μιλήσεις ευ, ευρωαγγλικά. Όχι, εγώ μιλάω δανοαγγλικά. Ντάνκης. Είναι δανέζικα και αγγλικά ένα μείγμα. Λοιπόν, έλεγα πάλι από την αρχή. Συμφωνώ απολύτως με τον Παλτσάκη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν εξαιρετική η ηγεσία σου και στην αντιπροσωπή μου. Πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις λοιπόν στις αρμόδιες αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το περιβάλλον, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, οδηγία για τον υδροφόρο ορίζοντα, η οδηγία για την Natura 2000 παραβιάζονται εδώ όπως είναι προφανές. Και επίση υπάρχει και η σύμβαση του όρου για την ενημέρωση και αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γερμανία την ίδια και διάφοροι αναφέρονται ισχυρίζονται ότι δεν είχαν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες. Και κάτι άλλο για το οποίο ανησυχώ βαθύτατα. Όλοι αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από τον άνθρακα και ο λιγνίτης είναι ο χειρότερος άνθρακας με διαφορά. και καταστρέφουμε το τοπίο γιατί η εξόρυξη γίνεται σε ανοιχτά ορυχεία, σε ε, στρώματα και καταστρέφει τα πάντα και το τοπίο και το περιβάλλον. Και κανείς από ό,τι φαίνεται μεταξύ των αρχών ε, δεν σκέφτεται το μέλλον. Όταν συζητούμε για νέες θέσεις απασχόλησης, αντί να σκεφτούμε πώς θα περάσουμε στις αηφόρες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτή. Έχουν εκεί πέρα κάτι ανανεώσιμες, αλλά πολύ ε, αποσπασματικά. Ε, τι γίνεται με εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν είναι καθόλου στην ημερήσια διάταξη. Ε, και είναι πολλές θέσεις απασχόλησης, ε, είναι όριμες οι συνθήκε για να μεταβούμε σε αυτή ε, την παραγωγή ενέργειας και αυτό δεν μπορεί να μετακατασταθεί ως βιομηχανία. Υπάρχει και κοινή ενεργειακή πολιτική που μιλάει για ενεργειακή απόδοση και για εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή γρήγορα μπορεί να περάσουν σε μια σύγχρονη παραγωγή αηφόρο Μα έλεγαν συνέχεια για το σοκ που πάθανε με την επανένωση το 90 και το σοκ που πάθανε το 2000 που χάσανε θέσει εργασία. Προφανώς. Αλλά θα τα ξαναβρούν μπροστά τους αυτά τα σοκ εάν δεν ε, προετοιμαστούν για τις σύγχρονες εποχές, τη σύγχρονη τεχνολογία και τον σύγχρονο ανταγωνισμό. Επανειλημμένα το είπαμε και οι απαντήσει ήταν ε, πάρα πολύ ασαφείς και καθόλου στραμμένες προς το μέλλον. Αυτό πραγματικά με ανησυχεί. Αυτός ο λιγνίτης, ακόμα και με την τελευταία τεχνολογία, είναι πολύ βρώμικο πράγμα. Μπορεί να αλλάξει τεχνολογία. Το υλικό δεν αλλάζει. Πραγματικά καταστρέφει το τοπίο αυτός ο τρόπος εξόρεξης. Αυτό ήθελα να πω. Καλό ήταν που πήγαμε Άλλη φορά μήπω να κάνουμε και καμιά δημόσια συνεδρίαση με κοινό για να ακούει ο κόσμος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί και ασχολείται. Εγώ φταίω, θα έπρεπε να το είχα ζητήσει στο πρόγραμμα, γιατί το έχω δει σε άλλε αντιπροσωπείε και άλλε αποστολέ. Είναι καλή ιδέα καμιά φορά να ακούν οι πολίτε ότι είμαστε εκεί και ενδιαφερόμαστε, ακούμε και ανησυχούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω το εξή ότι νομίζω δεν έχει κανένα νόημα να στείλουμε τώρα επιστολή στη γερμανική κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει καταρχήν κυβέρνηση. Ε, θα εξετάσουμε την ε, άνοιξη, την ε, έκθεση της Επιτροπής που θα έχει μεταβεί επιτόπου, όταν ελπίζουμε τότε να υπάρχει κυβέρνηση. Έχω άλλο έναν ομιλητή στον κατάλογο, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντανούκα. Και εγώ ήμουνα συμμετείχα σε αυτή την επιτροπή που μετέβη επιτόπου. Να ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Τσάκη, πολύ καλή η δική του η δουλειά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ε, όλη αυτή η υποστολή. Επικεφαλής βέβαια ήταν ο κύριος Τσάκη. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν η Μαργκρίτε και ο κύριος Τσάκη. Απλά θέλω να επισημάνω ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας εξετάσαμε κι άλλη μία αναφορά η οποία ε, προέρχεται από το Βερολίνο και ε, αφορά την μόλυνση του ποταμού Σπρέ που προέρχεται η ρήπανση αυτή από τα λιγνητορυχεία, ε, η αναφορά εκκρεμή ακόμα, το πρόβλημα της ρήπανσης σε όλη αυτή την περιοχή από το Πότσταμ μέχρι τη Δρέσδη, το όλο θέμα πράγματι υπάρχει και δεν έχει επιληθεί. Ε, πρέπει να σας πω εξεπλάγει και για το ε, Πώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα τη ε, γερμανικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι πρέπει να καταθέσουμε ε, σύσταση στην έκθεσή μας για τη νέα γερμανική κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και για τις τοπικές κυβερνήσεις και έτσι νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την έκθεση της Επιτροπής. Η Μάργαρετ, πάρα πολύ σύντομα να πω ότι η Τατιάνα φεύγει φεύγει. επιστρέφει στη Λετωνία για να συνεχίσει τη δουλειά της ε, με τις ε, μειονότητες. Αυτή ήταν η τελευταία της παρέμβαση ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συμμετοχή της. Ε, πρέπει να ευχαριστήσουμε την ε, Τατιάνα για τη δουλειά που έχει κάνει και έχει προσφέρει τη δική της άποψη σε αυτήν την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους σας ε, για το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε. Νομίζω ο αντικαταστάτης μου ή η αντικαταστάτριά μου θα συνεχίσει τη δουλειά μου. Δεν ήξερα, Τατιάνα, ότι επιστρέφεις στην πατρίδα σου. Ε, σου εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, τα καλύτερα, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το να συνεργαστούμε μαζί σου. και έχουμε βέβαια και ένα πρόβλημα διαφθοράς σε σχέση με τις μειονότητες, θα λυθεί και αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η παρουσία σε μελετής για τα σχέδια διαχείριση πληθυσμών μεγάλων σαρκοφάγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στου εμπειρογνώμονε Ντουάρτε Καντέτα Νταρόχα Περέιρα ε, και στην κυρία Μαρία Ντίας Πίντο Φερέιρα. Παρακαλώ. Uh, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας παρουσιάσω το έργο μας για τα σχέδια διαχείρισης μεγάλων σαρκοφάγων ε, στη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση ε, για να σας ε, αναφέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε για τα ζώα. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται σε τέσσερα είδη, τα οποία είναι ενδυμικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καφέ αρκούδα, ο λίγκας ευρασίας, ο λίκος και ο αδιφάγος. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για έτοιμα ε, κάποιας αναφοράς και για να σας παρουσιάσουμε το νομικό πλαίσιο για τα μεγάλα σαρκοφάγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνθήκες ε, παρέκκλησης ε, αυτών των νομικών μέσων, να σας παρουσιάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για τη μίεση των προβλημάτων μεταξύ των ειδών αυτών και των τοπικών κοινοτήτων και να κάνουμε και συστάσεις προς τους ηθήνοντες. Το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα μεγάλα σαρκοφάγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίστηκε για πρώτη φορά το 1979 με την ε, σύμβαση της Βέρνης ε, και μετά είχαμε την οδηγία Habitat ε, το 1992 που είναι το νομικό μέσο το οποίο ρυθμίζει την προστασία των μεγάλων θηλαστικών σαρκοφάγων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Επιπλέον αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ειδική νομοθεσία για την προστασία των μεγάλων σαρκοφάγων. Η καφέ Αρκούδα όπως βλέπετε βρίσκεται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, στην Ανατολική Ευρώπη και υπάρχει και μικρός πληθυσμός κατακαιρματισμένος στην Ιβυρική Χερσόνησο και στην Ιταλία. Είναι προστατευόμενο είδος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείται ότι είναι σε ανεπαρκή ή ακατάλληλη κατάσταση, στη, ανεπαρκή κατάσταση στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ε, σχετίζονται ε, κυρίως και με την ερμηνεία και ε, κάνουν ζημιές σε μελισσοκομικές εκτάσεις και φυσικά καταναλώνουν τρόφιμα και επιτίθενται σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν ε, και θανατηφόρες περιπτώσεις ε, και υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης ε, και κάνουν και επιθέσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ο Λίγκα της Ευρασίας εμφανίζεται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, σε ανατολικές χώρες και στην κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την Εστονία, τη Λετωνία και τη Φιλανδία το καθεστώς συντήρησης θεωρείται κακό ή ανεπαρκές στις περισσότερες χώρες μέλη. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι ίσονα σημασία σε σχέση με άλλα μεγαλύτερα σαρκοφάγα και κυρίως ε, σχετίζονται με επιθέσεις σε πρόβατα. Ε, η διαχείριση ε, μέσω θανάτωσης από, ε, δείχθηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική για να μειώσει τα προβλήματα και τις ε, επιθέσεις σε πρόβατα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη συνύπαρξη με το άλλο μεγάλο θηλαστικό, τον αδιφάγο και τις βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να είναι η χρήση προληπτικών μέτρων όπως για παράδειγμα φύλακες για τα κοπάδια ε, φράχτες ε, ή άλλες μορφές προστασίας. Ο λύκος είναι το πιο διαδεδομένο σαρκοφάγος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως βλέπετε εμφανίζεται σε διάφορα κράτη-μέλη. Είναι ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος, εκτός από την Εστονία, τη Λετονία, ε, την Φιλανδική έκταση στην Πολωνία, και στην Ισπανία, στα βόρεια τμήματα. Θεωρείται ότι είναι σε κακή ανεπαρκή κατάσταση σε 11 από τις 17 χώρες στις οποίες εμφανίζεται το είδος. Ε, υπάρχουν προβλήματα κυρίως ε, με επιθέσεις σε κοπάδια και ε, υπάρχει και ανταγωνισμός στο κυνήγι με τους κυνηγούς. Ε, η διαχείριση μέσω θανάτωσης επίσης δεν ήταν αποτελεσματική ε, γιατί δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με το είδος αυτό και δεν μείωσαν και τις συνέπειες ε, για τις ζημιές στα κοπάδια. Ε, οι βέλτιστες πρακτικές συνύπαρξης είναι η χρήση προληπτικών μέτρων όπως αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως και ιδίως ε, ε, βελτιώσεις για την ε, αποδοχή των λύκων. Αυτό μπορεί να γίνει με εκστρατεία ενημέρωση, συμμετέχει ενδιαφερομένων όπως ομάδες κυνηγών, γεωργών και στήριξη προς αυτές τις ομάδες. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε και ε, τα άγρια θυράματα σε περιοχές τις οποίες ε, δεν υπάρχουν. Και τέλος, ε, το τελευταίο είδος είναι ο αντιφάγος. Πρόκειται για ένα είδος το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μόνο στις σκανδιναβικές χώρες. Έχει ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης μόνο για τις περιοχές Τη Φιλανδία, που έχουν βιοκλιματικές συνθήκες αντίστοιχες με τις Άλπες. Είναι δηλαδή μια ορεινή ε, περιοχή. Ε, θεωρείται ανεπαρκές ε, ή ανύπαρκτη η κατάσταση για το είδος και τα προβλήματα είναι ίσονο σημασία, διότι εμφανίζεται σε πολύ μικρό τμήμα της Ευρώπης και συνήθω σχετίζεται με επιθέσεις σε κοπάδια προβάτων ή ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα αποζημιώσεων, αυτό προτείνεται και η διαχείριση μέσω θανάτωσης επίσης αποδείχθηκε ότι δεν είναι αποτελεσματική για να μειώσει την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τις επιθέσεις στα κοπάτια. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες ε, για παρεκκλήσεις βάσει της οδηγίας Habitat, εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά την έννοια της παρέκκλησης. Η παρέκκληση είναι μια εξαίρεση για την ε, προστασία ενός συγκεκριμένου είδους. Συνήθως μπορούμε να άρουμε την ε, παρέκκληση μέσω θανάτωση σε κάποιον ε, άγριο πληθυσμό και πρέπει να κατανοήσουμε και τι σημαίνει ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, το οποίο από εδώ και πέρα θα αναφέρουμε τα αρχικά του, FCS. Το FCS σημαίνει ότι ε, το είδος διατηρείται, είναι βιώσιμο, ζει στο φυσικό του περιβάλλον, δεν μειώνονται τα αποθέματά του και δεν προβλέπεται μείωση για το εγγύς μέλλον ε, υπάρχει ε, επαρκής ε, παρουσία του είδους ε, στη συγκεκριμένη περιοχή κατοικίας του. Τώρα, στο παράρτημα 4 της οδηγίας Habitat μπορεί να υπάρχουν παρεκκλήσεις μόνο όταν δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές εναλλακτικέ λύσεις και αν αυτό δεν είναι εις βάρος του καθεστώτος διατήρησης των ζών. Ε, βάσει του παραρτήματος 5 της οδηγία ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε παρεκκλήσει μόνο όταν θεωρούνται απαραίτητε ε, και η αεάνη απομάκρυνση των ζώων και η εκμετάλλευσή τους αφορά και είναι με βάση το FCS. Όσον αφορά τα, την εκμετάλλευση των μεγάλων σαρκοφάγων, εδώ θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην Ευρώπη και τα τέσσερα αυτά είδη δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης για υποστήριξη, δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ε, και επομένως οι δράσεις αυτές δεν συνάδουν με το πνεύμα της οδηγίας Habitat ε, και με τις απαιτήσει ε, της οδηγίας. Δεν είναι συμβατά με τη διατήρηση ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης και επειδή παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη γεωγραφική ποικιλομορφία, όλα αυτά τα είδη μπορεί να εμφανιστούν και να δείξουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ε, σαρκοφάγων. Και πρέπει να δούμε τι μπορούν να κάνουν αυτά τα τέσσερα είδη και να τα λάβουμε δεόντως υπόψη. Ένας από τους πιο κοινούς λόγους για τους οποίους τα κράτη-μέλη ζητούν παρεκκλήσεις είναι γιατί έχει μειωθεί... Ε, λόγω της παρουσίας των σαρκοφάγων αυτών ε, ο αριθμός των κοπαδιών. Αλλά ε, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν και αντίστροφα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ για παράδειγμα έχουμε ε, μία μελέτη για τη σχέση λύκων και μείωση του αριθμού των κοπαδιών και εδώ βλέπουμε στα αριστερά ένα διάγραμμα που είναι το αναμενόμενο λόγω της αναλογίας απώλειας με τη μείωση των λύκων αλλά αυτό το οποίο συνέβη στην πραγματικότητα είναι αυτό που έχουμε στα δεξιά στο διάγραμμα. Εδώ βλέπουμε ο αριθμός των απολειών ουσιαστικά αυξήθηκε ε, όσο ταυτόχρονα θανατώνονταν ή απομακρύνονταν οι λύκοι. Ε, μετά λοιπόν από ε, την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού λύκων τελικά ε, μειώθηκαν οι απώλειες στα κοπάδια αλλά ο αριθμός ε, των ε, λύκων που απομακρύνθηκαν δεν συνάδει με το καθεστώς FCS ε, και δεν συνάδει και με το πνεύμα της οδηγίας Habitat. Ένας άλλος κοινός λόγος για να ζητήσουμε διαχείριση μέσω θανάτωσης είναι για να βελτιώσουμε ε, την ε, ε, ανοχή των μεγάλων σαρκοφάγων, αλλά οι μελέτες έχουν καταδείξει ότι μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό του λαθροκυνηγιού και φυσικά αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και όλα τα προβλήματα που αφορούν κοινωνικές αντιλήψεις και προβλήματα. Ένα άλλο λόγο για να ζητήσουμε διαχείριση μέσω θανάτηση είναι για να ελέγξουμε τον αριθμό του πληθυσμού. Αλλά όλα αυτά τα είδη έχουν μοναδικά βιολογικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ε, αργή διαδικασία αναπαραγωγή ε, και επομένω υπάρχει έλεγχο στον αριθμό του. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε εμεί έλεγχο στον αριθμό του πληθυσμού μέσω θανάτωση των ζώων. Και επίση ε, αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να διαταραχθούν πάρα πολύ με διαχείριση μέσω θανάτωση. Ε, σε συμπέρασμα, για να δώσουμε και κάποιες συστάσεις, προτείνουμε ε, να χρησιμοποιούνται προληπτικών μέτρα διότι είναι τα πιο αποτελεσματικά, τα πιο δίκαια και τα πιο ε, ε, εύκολα να εφαρμόσουμε για να μειώσουμε τα ε, προβλήματα από τη μείωση των κοπαδιών. Για παράδειγμα, να υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα. Αυτό είναι χρήσιμο εργαλείο και θα έπρεπε να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο. Προγράμματα αποζημίωση επίση, τα οποία θα πρέπει να είναι δίκαια και να υποστηρίζονται και από την έγκριση προληπτικών μέτρων για παράδειγμα εδώ ε, διάφορες μέθοδοι όπως για παράδειγμα φύλακες για τα κοπάδια και άλλα μη παραβατικά παραδοσιακά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Ε, παρεκκλήσεις ε, οι οποίες αφορούν τον έλεγχο των ειδών και περιλαμβάνονται στο παράδειγμα 4 και 5 πριν εφαρμοστούν θα πρέπει να αξιολογηθούν πάρα πολύ καλά. Η διαχείριση των μεγάλων ε, σαρκοφάγων θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές αρχές ε, μέσω μιας στρατηγικής υποστήριξης, ενημέρωσης ε, και διαφάνειας για τους διαφόρους ενδιαφερομένους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας, να έχουμε μια νέα προσέγγιση οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές της επιστήμης δεν θα πρέπει απλώς να θεωρούνται ότι είναι το ενδιαφέρον κάποιο ακόμα, αλλά θα πρέπει να αποτελούν την πηξίδα που θα ε, ε λαμβάνουμε υπόψη μας και αν ε, διαβουλευτούμε και όλους τους ε, υπόλοιπους ενδιαφερομένους, κυνηγούς, αγρότες κλπ, θα πρέπει πρώτα να παίρνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της επιστήμης. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσουν την οικονομική στήριξη για την επιστημονική έρευνα για την πρόληψη των ζημιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η στήριξη και η έρευνα θα πρέπει να γίνεται πριν ληφθούν πρακτικά μέτρα ε, επιτόπου, διότι εάν η έρευνα γίνει εκ των προτέρων, πιστεύουμε ότι τα μέτρα θα είναι ε, πολύ καλύτερα και θα βελτιωθούν περισσότερο στο μέλλον. Και τέλος, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πίες, για παράδειγμα, κάτι πολύ απλό που γίνεται, αν δεν αποδειχθεί επιστημονικά ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί ένα ζώο από το φυσικό του περιβάλλον, τότε δεν... Okay. Oh, το συνάδελφο, βλέπετε τα ονόματα εδώ ε, και είναι πολύ, ε, πολύτιμη η μελέτη πραγματικά. Τουλάχιστον μπορούμε να εμπνευστούμε πολύ από εμά και να βρούμε και στρατηγικέ εκεί για να καταπολεμήσουμε ε, κάμια-δυο στρεβλές αντιλήψεις στον κόσμο. Θα δώσω το λόγο με χαρά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να, σας ευχαριστώ πολύ. Λύσεις. Το θέμα αυτό απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους να συμβιλιώσουν την διατήρηση αυτών των ειδών με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού για σας. Κάναμε έναν έλεγχο ε, της νομοθεσίας ε, κατά πόσο ανταποκρίνεται και είναι η κατάλληλη. Απεδείχθη κατάλληλη. Ε, βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει και χρειάζεται δουλειά είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας. Η νομοθεσία είναι καλή. Έχουμε ένα πρόγραμμα δράση από τα μέτρα που περιλαμβάνονται αφορά την ενημέρωση και την προώθηση των καθοδηγητικών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία και διατήρηση των ειδών. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή ξεκαθαρίζουμε ποια είναι η νομοθεσία και πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε. Το δεύτερο, είχαμε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα και έχουμε και τρεις νέες περιφερειακές πλατφόρμες ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα από αυτά. Και στόχος είναι πάντα η προώθηση, η προαγωγή του διαλόγου και αν στη μελέτη, όπως ακούσαμε, έχουμε την οδηγία Habitat για τους οικοτόπους που επιτρέπει να γίνονται παρεκκλήσεις για μεγάλα σαρκοφάγα υπό ορισμένους ε, όρους ε, με ε, επιλεκτική θανάτωση. Ε, αλλά υπό όρου Και το λέει και η μελέτη. Ε, τη μελέτη την ε, επεξεργάζομαστε αυτόν τον καιρό και θα τη συμπεριλάβουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνέχεια νέε μελέτε, θα τη δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μαντσελέζη πρώτος. Μαντσελέζη. Πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συντάκτες της έκθεσης και της μελέτης. Συμφωνώ πολύ που αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι και για την εμπορευματοποίησή του. Πρόσφατα παρουσιάστηκε η μελέτη αυτή τη Βρυξέλλη. Επιτέλου έχουμε μια μελέτη που βασίζεται σε επιστημονικέ αρχέ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών. Αυτή τη Βρυξέλλη. Επιτέλου έχουμε μια μελέτη που βασίζεται σε επιστημονικέ αρχέ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα στο πνεύμα των Ευρωπαϊκών νόμων και αυτό εκ των Θα ήθελα εδώ να τονίσω μερικά σημεία. Πρώτον, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει κανένα νόημα να σκοτώνουμε το λύκο και να κυνηγάμε το λύκο. Δεν, δεν βοηθάει. Το έχουμε δει στην Ισπανία επανειλημμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για, ε, να τηρείται η νομοθεσία και από εκεί ε, θα ξεκινήσει και η λύση των προβλημάτων. Αν έχουμε αντισταθμιστικές πληρωμές, αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν πάντα και με μέτρα και τα μεγάλα σαρκοφάγα μάλλον και το λύκο. Αλλά θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ευρωπαϊκό μας ε, έργο και να τους βοηθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τις χώρες να αποφασίζουν η μία να κυνηγάει το λύκο, η άλλη να κάνει ε, εξόντωση ε, της επιλεκτική όχι, πραγματικά στην πρόληψη, στην εκπαίδευση και στην ύπαρξη και στη συμβίωση με βάση επιστημονικά στοιχεία. Δύο προτάσεις θέλω να κάνω. Μία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πραγματικά θα ήθελα να ε, επέμβεται στην Ισπανία, έχοντα διαβάσει αυτή τη μελέτη, γιατί αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μου σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με αυτά που ακούσαμε στον χωρό μα που έχουμε μεγάλα σαρκοφάγα. Και σα παρακαλώ στην Ισπανία οπωσδήποτε να το στείλουμε για το λύκο, διότι πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουν και τη φωνή της λογικής και τη φωνή της επιστήμης και τη φωνή της κοινή λογικής, σε πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέταγιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε ότι στην Επιτροπή Αναφορών ε, έχουμε πάρει αρκετές αναφορές ε, για το λίκαλα, το θέμα της διαχείρισης του προβλήματος του λύκου. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα. Στη Γερμανία υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η λύκη, αυτή είναι μια καλή είδηση ότι οι λύκοι κάπως έχουν εγκατασταθεί στη χώρα. Και καλό είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως ε, πρέπει να δει κανείς και τι συμβαίνει με τις τοπικές, τις τοπικές κοινωνίες όλο και περισσότερο περιορίζεται έναντι των λύκων. Όσον αφορά τη διαχείριση του προβλήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αλλάξει ορισμένα πράγματα να τα βελτιώσει. Ξέρετε κατά τη δική μου άποψη και στη Γερμανία έχουν γίνει προβλήματα. Δηλαδή υπήρξε κάποια διαχείριση του προβλήματος του λύκου, οι λύκοι. Αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον δεν έγινε σαφές στους πολίτες. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και πολιτικό το πρόβλημα. Ε, βλέπει κανείς ε, ότι οι πολίτες έχουν ε, λιγάκι ριζοσπαστικοποιηθεί και πολιτικά γιατί θεωρούν ότι τους έχουν ζημίωση. Είμαστε ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατάργησε τον κανισμό de διότι μπορεί σε επίπεδο χώρας να μην ζημίωση. Είμαστε ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατάργησε τον κανισμό de διότι μπορεί σε επίπεδο χώρας να μην αποτελεσματικά τα προστατευτικά ε, μέτρα. Στο παράρτημα αναφέρεται ότι αν παραδείγματο χάρη περνάνε ολόκληρε εβδομάδε μέχρι κοινωνία, αν το κάνει πρέπει να απομακρυνθεί και αν αυτό διαρκεί εβδομάδε δεν εξηγείται εύκολα. Θέλω λοιπόν να πω το εξή, ότι χρειασέξουμε. Ε, πρέπει να σα πω ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά, πολύ στραβά καλό το παράδειγμα, αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί νομίζω ότι παραδείγματος χάρη, αν πάει κανείς προς τα πάνω, ε, προς, την, προς τις ακτές, εκεί έχουμε τις θύνες ε, Παραδείγματο χάρη, αν πάει κανεί προς τα πάνω, προ ε, τι προς ακτές, εκεί έχουμε τι θύνες ε, και τα πρόβατα και αν πάνε εκεί οι λύκοι, τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Προστατευτικά μέτρα δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Από την άλλη όμως ε, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και νομίζω ότι δεν πρέπει να καταλήγουμε στο ότι κυνηγάμε τα πρόβατα πριν μπούμε σε ένα επικίνδυνο δάσος. Δεν είναι σωστή αυτή η λογική. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβάσει τις αναφορές και τις δύο. Να διαβάσει αυτές που λένε ότι κάνουμε πολύ λίγα για το λύκο, αλλά να διαβάσουν και τις άλλες που λένε ότι κάνουμε πάρα πολλά για το λύκο. Κάπου να βρεθεί μια ισορροπία και εντωμεταξύ ε, χρειαζόμαστε και κάποιες ε, λύσεις ε, που να ικανοποιούν και τους ανθρώπους και τα ζώα, τους λύκους. Πολύ σημαντικό. Τώρα στα Δανέζικα θα τα πεις για τους λύκους, Μάργαρετ. Κυρία Όκεν. Ναι. Καμιά φορά μπορεί να ακούνε και δανείοι, οπότε δεν πρέπει να μιλάω αγγλικά εγώ. Ε, γινόταν κάποια φασαρία και ρωτήσαμε τους ε, Ρώσους τι έγινε και είπανε ότι είχαν εξαλείψει τα κουνούπια από το Σότσι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι, πώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήταν καταστροφή από πλευράς βιοπικιλότητας. Και ο Λύκος είναι δώρο για μας. Όπου ε, φεύγουν κάποια ζώα, υπάρχουν ξέρω, κάποια ελάφια που φεύγουν, έρχονται άλλα ζώα. Έτσι, όπου ε, φεύγουν κάποια ζώα, υπάρχουν ξέρω, κάποια ελάφια που φεύγουν, έρχονται άλλα ζώα, έτσι να καταστρέφεται και να υποχωρεί ε, με την εξαφάνιση των ειδών. Και ο λύκος ανήκει στη βιοπικιλότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα πρόβατα τώρα. Στο παρε... Και να φυλάνε το κοπάδι. Και αποθαρρύνουν τους λύκους. Και εμάς μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους ανθρώπους που παρουσίασαν σήμερα αυτή τη μελέτη. Πολύ σημαντικά γιατί όπω και ο συνάδελφο Ματσελέ των μελών. Και αυτό ισχύει και για την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία είναι μία από τις χώρες όπου δυστυχώ, η Ιταλία ε, αναθεωρεί λιγάκι το εθνικό τη πρόγραμμα για το λύκο. Από το 1961 είχε απαγορευτεί το κυνήγι, τώρα όμως σκέφτονται να μελέτη του συναδέλφου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και ιδιαίτερα το να δοθούν αυτές τις πληροφορίες στα κράτη-μέλη για να αποφύγουμε έτσι ώστε να επανέλθει το ενδεχόμενο του κυνηγιού που τώρα πραγματικά δεν μπορεί να εφίσταται τέτοιου. Υπάρχει η ρήπανση, η, ε, η διάβρωση των υδάτων. Ε, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα στις ε, πόλεις μας με τεράστιες ζημιές στο οικοσύστημα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ απευθύνομαι στην Πρόεδρο να στηρίξει την μελέτη. Να το προσέξουμε πάρα πολύ και να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους να συζητούν, να κατεβάσουν λίγο τα όπλα τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη, αυτό είναι το βασικό, που στι μόνιμες αντιπροσωπείες το διαβιβάζουν αρμοδίω. χώρε του. στις χώρες τους. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το να στέλνει από εδώ κάτι σκητά με 18 υπογραφέ, σχετικά με την εικαζόμενη ανεπαρχική εφαρμογή της οδηγία πλαισίου περί υδάτων στο κρατήδιο τη κάτω Σαξονία. Ε, είναι το εξής. Ε, πρόκειται ε, για τα ορυχεία αλάτου στην περιοχή βελτιώσει τις πρακτικές τους επί του θέματος ε, και από ό,τι φαίνεται έχουν και ένα master plan ε, για την παραγωγή άλατος. Αυτό είναι χρήσιμο για να το δηλαδή ακόμα δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα συγκεκριμένο που να ε, μπορεί να αποτελεί κάποια παραβίαση. τόσο η οδηγία περί πολύ πρόωρη φάση φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ ωραία, λέει η πρόεδρος. Από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοι εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που να θέλει να λάβει το λόγο επ' αυτού του θέματος. Από ό,τι βλέπω όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα δεν λειτουργήσε η κάρτα μου για να ψηφίσω. Ήλπιζε λοιπόν τουλάχιστον θα λειτουργήσει το μικρόφωνο μου και να που Έχω λοιπόν μπροστά μου κάποια έγγραφα όπου αναφέρεται ότι για το πρόγραμμα αυτό ε, υπάρχει και κρεμεί μελέτη συμβατότητας με το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα προκύψει ακόμα. Ως εκ τούτου εμείς θεωρούμε ότι η αναφορά αυτή μπορεί να κλείσει. Πράγματι και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσει το θέμα και να αναφέρουμε ύβρομενο θέμα το 2097 ε, σχετικά με τις επιβλαβείς δηλαδή επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία που προκαλούνται από μια γραμμή υψηλή τάσης στη Βόρεια Πορτογαλία. Ε, πρέπει να σας πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Καταγγελία η οποία επιβλήθη τον Οκτώβριο του 2014 μέσω Τη Άννα Μιράντα και τη Μαρίζα Αματίας. Η Άννα Μιράντα ήταν τότε ευρωβουλευτής ε, και τις ευχαριστούμε και τις δύο και αφορά το ε, πρόγραμμα υψηλής τάσης, ε, συγκεκριμένα τον αριθμό πτώσης της τάσης. Πέσανε 7 πυλώνες. Το 2013 έγινε μια μελέτη και σύμφωνα με αυτήν ε, αποφασίστηκε η κατασκευή. Σημεία αυτά είναι τα πιο ε, ευαίσθητα σημεία της ε, γραμμής. Αυτή η γραμμή υψηλής τάσης θα περνάει από την περιοχή της Βαλίνιας οι πόστες ε, και ε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο στοιχείο της ε, γραμμής και θα περάσει κοντά από κατοικίες και θα δημιουργήσει προβλήματα σε τέσσερις περιπτώσεις και θα υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν θα υπάρχει ηλεκτροδότηση στις κατοικίες των περίκων και γι' αυτό θα υπάρχει πρόβλημα και με τα ηλεκτρονικά πεδία και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο ζητάμε τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση του 2008 ε, βάσει και τι οδηγίες που ζητούν ε, εγγυήσει ε, ασφαλείας γραμμή υψηλή τάσης. Μέχρι σήμερα προβλέπεται να... τι γίνεται, να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τους ε, περίοικους, διότι είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικίες ε, ε, και γι' αυτό ακριβώ το λόγο ζητάμε να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης στο πρόγραμμα αυτό και επίσης ζητούμε να επιλύσει το θέμα της ολοκλήρωσης του θέματος και να δούμε τι γίνεται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ε, μεταξύ της περιοχής αυτής και των ε, πορτογαλικών συνόρων. Αυτή η κατασκευή της γραμμής υψηλής τάσης βρίσκεται στη διαδικασία. Γίνεται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ε, μεταξύ της περιοχής αυτής και των πορτογαλικών συνόρων. Αυτή η κατασκευή της γραμμής υψηλής τάσης βρίσκεται στη διαδικασία προκειμένου να ε, ολοκληρώσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά η ισχύουσα νομοθεσία σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει ότι αφή στιγμή ξεκινήσει η διαδικασία της τεχνικής εξέτησης ε, το 2014 μπορεί μέχρι και σήμερα το 2018 να μην έχει ολοκληρωθεί. Τρία χρόνια και δέκα μήνες δηλαδή από τότε που ξεκίνησε και ε, εκρεμεί η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Ένωσή μας ε, θεωρεί ότι οι προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται βάσει της ε, ε, νομοθεσίας θα πρέπει να τηρούνται και επομένως θεωρούνται ότι εδώ δεν υπάρχει συμμόρφωση βάσει και της νομοθεσίας περί εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχουν αρκετές αναφορές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Ζητάμε ενημέρωση για την ε, ε, υποβολή της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παρουσιάστηκε ε, στο Δημαρχείο της περιοχής το Νοέμβριο του 2017 γιατί σε εκείνο το στάδιο μελετών ξεκίνησαν και οι συμβάσεις με τους Δήμους και έγιναν συνεδριάσεις με τους εργολάβους και έγιναν και διάφορες μελέτες επιτόπου. Το πρόβλημα είναι ότι το έγγραφο αυτό χάθηκε και δεν ε, έχει καταχωρηθεί. Και επομένως ε, δεν λήφθηκε υπόψη στο ε, στάδιο των διαβουλεύσεων και δεν μπόρεσε να ληφθεί υπόψη το έγγραφο. Επίσης, δεν έγινε γνωστό δημοσίως επειδή ακριβώς απολέστηκε και εμείς από πλευράς ε, της Ένωσής μας στείλαμε 14 επιστολές στο Υπουργείο Βιομηχανίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ζητώντας πληροφορίες, αλλά ε, η δυσκολία ήταν ότι τα Υπουργεία αυτά δεν μας απαντούν και ε, δεν μας λένε για την κατασκευή της γραμμής υψηλής τάσης, παρά το γεγονός ότι ξέρουν ότι υπάρχουν οι πληροφορίες. Επειδή λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό είναι έλλειψη σεβασμού ε, και δεν μας απάντησαν, καταγγείλαμε στον ε, ε, ε, Ισπανό διαμεσολαβητή το γεγονός και το 2017 ο Ισπανός διαμεσολαβητής απάντησε για δεύτερη φορά και θεώρησε ότι το Υπουργείο Βιομηχανίας ε, είναι ε, αδικαιολόγητο που δεν έδωσε απαντήσεις ε, και οι πληροφορίες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αιτιολογήσουν και κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει μια εναλλακτική γραμμή. Ακόμα και σήμερα όμως η Ένωσή μας το Φεβρουάριο του 2018 δεν έχει λάβει απάντηση από το Υπουργείο. και δεν έχουμε λάβει στοιχεία για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη και δεν έχουμε και προηγούμενη τεκμηρίωση. Τώρα, ε, για να τηρεί την ομοθεσία για την ε, αρχή της προφύλαξης και την ασφάλεια στη γραμμή υψηλή τάση, ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών να διατηρήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά και ζητάμε τη στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό την ελάχιστη απόσταση των ε, γραμμών υψηλή τάσεω από κατοικημένε περιοχέ. Άρα, αυτή την ελάχιστη απόσταση των ε, γραμμών υψηλή τάσεω από κατοικημένε περιοχέ. Άρα, από την άλλη, όπω είπα και αναφέρουσε, βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το έργο. Ακόμα δεν έχει δοθεί καμία άδεια. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια τόσο πρώιμη φάση της διαδικασίας τελεστεί αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να το λόγο. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για την ε, παρουσίασή της. Υπάρχουν εδώ δύο πράγματα που ανησυχούν σε αυτό το μεγάλο έργο σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μας έδωσε καμία γραπτή εξήγηση σχετικά με την τεκμηρίωση του έργου, ε, στοιχεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ε, ε, στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στην ενημέρωση για την περιβαλλοντική νομοθεσία, σύμφωνα με τη σύμβαση του Όρχους. Να, να παραμείνει ανοιχτή ζητούμε εμεί η αναφορά, να ζητήσουμε πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η οδηγία δεν παραβιάζεται κατά την άποψή μας για την περιβαλλοντική μελέτη και για τις επιπτώσεις του έργου αυτού στην υγεία του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Αναφέροντες ή τις αναφέρουσες, έχω μία παρατήρηση να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν υπάρχει ακόμα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι όμως πρόβλημα, γιατί εδώ η μελέτη αυτή είναι ε, νοσιακό δίκαιο, έχει καθυστερήσει εδώ και κάποια χρόνια και δεν είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει αυτό ε, να είναι εθνικό θέμα, να απευθυνθείτε στα εθνικά δικαστήρια. Δεν είναι σωστό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει επανειλημμένα ότι το θέμα αυτό δεν μπορούμε να το αφήνουμε στα εθνικά δικαστήρια. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι σαν να λέμε σκασίλα μας. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πολύ σημαντική, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο και ε, δεν είναι ε, βέβαια σωστό εκ των υστέρων να λέμε ότι α, δεν το ξέραμε. Αυτό σημαίνει αρκετά συχνά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε να δουλεύουμε και είμαι σίγουρη ότι και αυτός δεν είναι και ο τρόπος που θέλει να δουλεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να είναι όμως διαφορετικά τα πράγματα ε, πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Να παραμείνει ε, το θέμα ανοιχτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόεδρο, η κυρία Ευχαριστώ και την αναφέρουσα. Καταρχάς, θέλω να πω το εξή. Πρώτον, θέλω να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την Επιτροπή μας να πω στις 8 Φεβρουαρίου του 2017 σε συνεδρίαση με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας μας είπαν ότι το αρχικό έργο είχε αλλάξει. Έκτοτε βρισκόμαστε συνεχώς σε άγνοια και προσπαθούμε να μάθουμε ποια είναι η νέα χάραξη της γραμμής υψηλής τάσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παραπέμπει στην Ισπανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Ισπανική κυβέρνηση έχει στα χέρια της το έργο. Τρεις φορές ήρθαμε σε επαφή με το αρμόδιο Ισπανικό Υπουργείο και μας αποκρύπτουν πληροφορίες και στους πολίτες που θίγονται γιατί περνάει από τα σπίτια του η γραμμή αλλά και σε εκείνους που ε, έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν όπως εγώ ως βουλευτής ας πούμε το η Ισπανική κυβέρνηση δεν απαντάει και τρίτη, στην τρίτη απάντηση με παραπέμπει στην Επιτροπή Αναφορών. Αποταθείτε, λέει, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μάθετε. Αυτά είναι απαράδεκτα. Και επίση παραβιάζεται το παράρτημα 6 στι οδηγίε για τη διαφάνεια και τη δημόσια διαβούλευση στον κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση 347 του 2013 που ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση για τους ιδιοκτήτες άνδρες και γυναίκες και για τους πολίτες άνδρες και γυναίκες που είναι περίοικοι. Επίσης λέει θα πρέπει να υπάρχει στο σελίδα του έργου που να ανταποκρίνεται με τα προαπαιτούμενα που αναφέρονται στο παράρτημα 6 του ε, και έχει αλλάξει η χάραξη της γραμμής. Ωραία. Πού θα πάει και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές αποκρύπτουν τις πληροφορίες αυτές. Οπότε, ε, τι ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτο, να υποχρεώσει την Ισπανική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με το λόγο παράρτημα και να γνωρίζουμε πού είναι η χάραξη, η νέα γραμμή, από πού θα περάσει. Δεύτερον, να παραμείνει προφανώς ανοιχτή η αναφορά. Και τρίτον, ε, συμφωνώ με τις προτάσεις που έκανε η αναφέρουσα και μεταξύ αυτών να εγκαταλειφθεί το έργο. Θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια Επιτροπή Αναφορών έτσι ε, ώστε αν μη τι άλλο να μάθουμε ποια είναι η νέα χάραξη της γραμμής. Αυτά που μας κάνουν απαράδεκτα. Ευχαριστώ και εγώ στα ισπανικά η κυρία Ματίας, ευχαριστώ και τις αναφέρουσες. Ε, σε αντίθεση με όλα αυτά που ακούω εδώ, δεν πρόκειται κάτι αφορά μόνο το Ισπανικό κράτο αλλά και την Πορτογαλία και τη Βόρεια Πορτογαλία. Ο υπό την έννοια αυτή, στα τέλη του 2014, η συνάδελφό μου Άννα Μιράντα και εγώ ε, κάναμε καταγγελία για τη χάραξη της γραμμής αυτής και να πούμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Το θέμα δεν αφορά μόνο την Ιβυρική, Χερσόνησο, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αναφέρθηκε επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τις συναδέλφους μου. Και να μην ξεχάσουμε ότι αυτά που συμβαίνουν αφορούν και τον πληθυσμό στη Βόρεια Πορτογαλία. Όπως ακούσαμε λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι να κλείσει η διαδικασία για λόγους μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μιλάμε για ευρωπαϊκή νομοθεσία και όχι εθνική. Να παραμείνει ανοιχτή αναφορά δεν ε, έχει τηρηθεί η οδηγία για την ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα. Ποτέ δεν κάλεσαν τους ενδιαφερόμενους για να διαβουλευθούν μαζί τους για αυτό το θέμα. Και αν έχω καταλάβει καλά την οδηγία αυτή, για να συμμορφώνουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καλούν σε δημόσια διαβούλευση τον πληθυσμό. Θέλω λοιπόν να πω ότι συμφωνώ με τις συναδέλφες που μίλησαν προηγουμένως και θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για όλα τα θέματα που ανέφεραν και οι βουλευτίνες και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση εδώ. Δεν μπορείτε να μας πείτε ότι εκκρεμεί μελέτη όλα είναι ανοιχτά, άρα να κλείσουμε την αναφορά. Πού να την κλείσουμε. Να περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει, να ε, συμμορφωθούν προς την οδηγία και μετά θα δούμε αν θα την... Ευχαριστώ. Βλέπουμε από την αναφορά, από τις παρεμβάσεις ε, και ε, τα διάφορα. Ευχαριστώ. Βλέπουμε από την αναφορά, από τις παρεμβάσεις ε, και τα διάφορα έγγραφα της τοπικής κυβέρνησης Γαλλικίας ε, και της Ισπανικής κυβέρνησης. Πρόκειται για διασύνδεση Ισπανίας-Πορτογαλίας στην επαρχία Ποντεβέδρα. Ε, ακόμα δεν έχει έρθει η μελέτη ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγώ μαθαίνω ότι χρειάζονται κάποιες πρώτερες μελέτες. Η Ισπανική ΔΕΗ, ο διαχειριστής του δικτύου μάλλον της Ισπανίας και της Πορτογαλίας είναι αρμόδιοι οι δύο ομόλογοι αυτοί, ενέχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντες, το Υπουργείο Γεωργίας, και Περιβάλλοντος, περιμένουν όλε τι προκαταρκτικέ εκθέσει και η Διεύθυνση και κυβερνήσει Πορτογαλίας και ε, Ισπανία και ο Δήμαρχο του Άρμπο και ο, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της τοπικής προσπαθούν να δουν ποια θα είναι η χάραξη που θα έχει συμφωνηθεί με όλου του περιοίκου, με όλο τον πληθυσμό. Γιατί το έργο αυτό από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό για να λυθούν και τα θέματα της ανανεώσιμης ενέργειας στην Γαλλικία και στην Πορτογαλία. Προφανώς είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να κλείσει η αναφορά, πρέπει να διευκρινιστούν όλα αυτά τα θέματα, οπότε και εγώ συμφωνώ και ε, ο αντίκτυπος να είναι όσο γίνεται μικρότερος για αυτό το στρατηγικό για την Γαλλική Ακλάδο. Ε, εφόσον δεν έχουμε όλα τα έγγραφα για τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν τη δείτε ή αν πλήρω. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά δημοσίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο που έχουμε ε, συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες να συμφωνούν τόσο πολύ. Είναι πραγματικά ευρύτατη συνένεση. Έχετε το λόγο για δύο-τρία λεπτάκια ακόμα. Βάλε, βάλε. Καλώς, καλώς. Ευχαριστώ. Έκλεισε το μικρόφωνο της ομιλήτρης μου. Στην Ολλανδία, στη στην Ελβετία και γυρίσαν οι άνθρωποι οι μετανάστες, μαζέψανε πέντε λεφτά να φτιάξουν ένα σπίτι. Και η πολιτική δεν είναι δίπλα από τα δικά του σπίτια που περνάει η γραμμή, περνάει από εμά που είμαστε αναλφάβητοι, οι εργάτες. Εγώ ε, πήγα σχολείο μέχρι τα 12, έχω πολιτήριο δημοτικό, γι' αυτό να ε, παρουσιάσουμε το μέλημα των κατοίκων της περιοχής και παρακαλούμε να μας υποστηρίξετε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Και για το θάρρος σας και για την ειλικρίνειά σας που τα λέτε πραγματικά έξω από τα δόντια. Και μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή Αναφορών να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ε, μια πλήρη μελέτη αντικτύπου περιβαλλοντικού, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εφόσον δεν έχει κατατεθεί αυτή η μελέτη, που είναι κρίσιμη. Και ως τότε ε, αφήνουμε ανοιχτή φυσικά την ε, αναφορά και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να ε, πανενοχλούμε ε, τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας φέρουν μια πλήρη μελέτη υπερβαλλοντικού αντικτύπου. Στο μεταξύ θα αποστείλουμε επιστολή ε, στις αρμόδιες αρχές και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία για να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουν ότι εμείς παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση. Και όπως είπα, ήδη, είπε και αναφέρουσα, αυτό το θέμα είναι ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό. Είναι διασυνοριακό μεταξύ δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά ανθρώπους. Και αφού υπάρχουν ανησυχίες από τους πολίτες, είναι δική μας ευθύνη σε τούτη εδώ την Επιτροπή να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Έχει αλλάξει το έργο από ό,τι ακούμε. Όπως το είπε και η κυρία Σάρα Ροντρίγκες. Έχει αλλάξει χάραξη από την αρχή την αρχική γραμμή, χρειαζόμαστε πλήρη ενημέρωση. Πώς έγιναν οι αλλαγές, προς ποια κατεύθυνση λοιπά Όλες τις λεπτομέρειες. Και έχοντας όλο την, αρχή, την αρχική γραμμή, χρειαζόμαστε πλήρη ενημέρωση. Πώς έγιναν οι αλλαγέ προ ποια κατεύθυνση λοιπά Όλες τις λεπτομέρειες. Και έχοντας όλα και Επιτροπή. Μάλιστα. Θαυμάσια. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Και εντωμεταξύ να σας ευχαριστήσω κυρία Κώστα που ήρθατε μέχρι εδώ και να σας ευχαριστήσω και για το πάθος σας για το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιη ότι η περιοχή από την οποία ήρθατε μέχρι εδώ και να σας ευχαριστήσω και για το πάθος σας για το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιη ότι η περιοχή από την οποία ε, καλή επάνωδο στη χώρα σας. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους και τώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη αναφορά που είναι η 328 με 12 υπογραφές σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων στη γεωργία, σε γεωργικά φάρμακα. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πανταχού παρούσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ σε φυτοφάρμακα λόγω της δουλειάς τους χωρίς να έχουν αναμερωθεί από τον εργοδότη τους και χωρίς να υπάρχει κατάλληλη προστασία. 8. Στις 26 Ιανουαρίου ο Επίτροπος έγραψε στους αναφέροντας επιβεβαιώνοντας ζητήσαμε να σταλούν οποιασδήποτε σχετικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Πληροφορίες που αφορούν την Οδηγία 2000 η Επιτροπή σχεδιάζει αυτόν τον έλεγχο, προγραμματίζει τον έλεγχο στη Γαλλία. Είναι βάση της οδηγιας 2928 η οποία καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα θεμάτων για τις ε, τρεις σημαντικές ε, πτυχές που αφορούν ε, τους αναφέροντας θα γίνει εξέταση. Αφορά την αποθήκευση και αγορά φυτοφαρμάκων, την εκπαίδευση αυτών που χρησιμοποιούν επαγγελματικά φυτοφάρμακα και συστήματα για συλλογή πληροφοριών για χρόνια και οξία δηλητηρίαση που σχετίζεται με την χρήση φυτοφαρμάκων. Και ο έλεγχος Είπαμε γίνεται βάση οδηγίας 2009-128, θα εξετάσει τα θέματα αυτά και οποιασδήποτε πληροφορίες ε, παρασχεθούν για τις οδηγίες 98-24 και 2004-37 θα ε, διαβιβαστούν στους συναδέλφους ε, από τη Γενική Διευθύνση Απασχόλησης. Όσον αφορά τον έλεγχο, είναι ένας έλεγχος ο οποίος θα γίνει ε, για τη χώρα, για τη Γαλλία και αξιολογή της Γαλλίας, ε, μία εκ των οποίων θα είναι η Βρετάνη και θα συναντήσουμε τις αρχές ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Της Γαλλίας, μία εκ των οποίων θα είναι η Βρετάνη και θα συναντήσουμε τις αρχές σε περιφερειακό επίπεδο. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα καταρτιστεί έκθεση και από εκεί και πέρα η έκθεση αυτή θα δοθεί στις αρμόδιες αρχές της χώρας προκειμένου να διευκρινίσουν ή να σχολιάσουν και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται η δημοσίευση να γίνει προς το τέλος του 2018, η δημοσίευση της έκθεσης. Λοιπόν, ε, όσον αφορά στην οδηγία 9824, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει αναφέρει ότι οι οδηγίες αυτές πρέπει να μεταφραστούν, να υιοθετηθούν σε εθνικό δίκαιο και στην περίπτωση αυτή αυτό αφορά τη Γαλλία. Πρόκειται βέβαια για μία μεμονωμένη περίπτωση που κατά κανόνα εμπίπτει σε εθνική δικαιοδοσία ε, εφόσον υποτίθεται ότι η Εθνική Νομοθεσία έχει υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία. Από αρχές σχετικά με την εφαρμογή των δύο προαναφερθεσών οδηγιών. Ως εκ τούτου αυτό είναι ένα θέμα που κατά κύριο λόγο εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Βεβαίως αν ε, μετά τον έλεγχο που αναφέρθηκε λάβουμε περισσότερα στοιχεία. Thank you very much. Very good. Margaret. Η Margaret. To the Commission and I've just suggested that we κά ε, και ζητήσαμε να εξετάσουν το θέμα και μετά η Κομισιόν να επανέλθει μετά και από μία επίσκεψη επιτόπου. Αυτά τα... Είναι ανοιχτό. Ωραία. Η Ελεονόρα όχι μένει ανοιχτό ε, και όταν θα υπάρχει Ελεονόρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ζητήσω αυτή η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή γιατί πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να λάβουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου που θα κάνει φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, και ακόμα και αν εξετάζεται για τα φυτοφάρμακα και την έγκριση των χημικών φαρμάκων ε, πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη μας γιατί προφανώς ε, ε, και αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο που κάνω, μέχρι σήμερα δεν έχουμε κατορθώσει να εγγυόμεθα ότι οι εγκεκριμένες χημικές ουσίες είναι πραγματικά ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία, ότι δεν προκαλούν ε, ζημιά στην ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλές ενώσεις, ε, θύματα από φυτοφάρμακα και πάρα πολλές μελέτες για αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, στην υγεία. Αναφέρομαι και στα κατάλοιπα, στα κατάλοιπα που υπάρχουν ε, στα ύδατα, στο έδαφος, ε, στα τρόφιμα. Ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όσον αφορά αυτό το θέμα, αυτή η αναφορά, για να υπάρξει περαιτέρω έλεγχος. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματικά ε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή τον έλεγχο που θα γίνει Μάιο-Ιούνιο. Και το, η τελική έκθεση θα γίνει προς το τέλος του, τους ε, καλή τύχη, εύχομαι. Ε, αναφορά στην 600 του Φελίτσε Σαρώνη Ε, αναφορά στην 600 του Φελίτσε Σαρώνη εξ ονόματος της Ασοτσιατσιόνε Αρέζε 5, συνοδευόμενη από 18 υπογραφέ κατά τη τροποποίηση σχεδίου αστική επέκταση εμπορικού ψυχαγωγικού χαρακτήρα μια πρώην βιομηχανική περιοχή. η Μικαέλα Πίβα ε, και ο Νταβίτ Κιόκολα είναι παρόντες ε, και θα ήθελα να σας δώσω... ...η οποία ήταν ε, βιομηχανική περιοχή και θα μετατραπεί σε περιοχή εμπορικού ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Εδώ έχουμε υγεία των πολιτών και τα συμπεράσματα. Η περιοχή ενδιαφέροντος της ε, περιοχής αυτής περιλαμβάνει τρεις δήμους, το Δήμο του Αρέζε, του Καρμπανιάτε και του, Μιλανάτε και του Λαϊνάτε που βρίσκονται ε, βορειοδυτικά του Μιλάνο και είναι μια περιοχή μεγάλης ε, ε κυκλοφορίας. Η περιοχή είναι περίπου 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι σε μια υπογραφή μεταξύ διαφόρων περιοχών της περιοχής για μετατροπή της βιομηχανικής αυτής περιοχής σε εμπορικού, ε, οικιστικού χαρακτήρα και ε, τριτογενούς. Ε, τον Απρίλιο του 2006, η εκλογική δέσμευση του 2012, που απέριψαν οι πολίτες ε, με την ψήφο τους. Εμπορικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή ε, ο εργολάβος από το 2016 έχει ζητήσει να αλλάξει 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, να προσθέσει μια μεγάλη ε, περιοχή που θα είναι ένα ε, επιπλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα, να προσθέσει μια μεγάλη περιοχή που θα είναι ένα επιπλέον στην Ευρώπη. οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, του ε, έργου, εάν διπλασιαστεί η έκταση του εμπορικού κέντρου σημαίνει ότι θα διπλασιαστεί και ο αριθμό των οχημάτων που θα προσπαθούν να φτάσουν στην περιοχή, στο εμπορικό κέντρο και επομένω θα υπάρχει επιπλέον ρήπανση τη περιοχή που ήδη είναι πάρα πολύ ε, κακή. Ε, είχαμε 76 ημέρε το 2016 πάνω από τα ε, επιτρεπόμενα όρια, το 2017 94 ημέρα και επομένω είμαστε πολύ πάνω από τι 35 ημέρε που προβλέπονται από την οδηγία 2008-50. Ε, τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι ε, προβλέπεται ε, κατάλληλη ποιότητα του αέρα λόγω του έργου. Υπάρχουν όμως κάποιες εχμές οι οποίες φτάνουν και στα 200 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο και επομένως πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και αύξηση κατά 55% της έκτασης του εμπορικού κέντρου σημαίνει ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη και σχετική τεκμηρίωση και στην Ιταλία καταγράφει επίσης ε, ε, επιδεινώνει χρόνιες καρδιαγιακέ παθήσεις και νεοπλασίε και μία μελέτη του 2013 υπολόγισε ότι σε βόμερα θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικέ συνέπειε και αν διπλασιαστεί η έκταση του εμπορικού κέντρου δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ζητάμε λοιπόν στον Ντάβιντε. Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μας ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έδωσε τη δυνατότητα, την Επιτροπή σας μάλλον, συγγνώμη, που μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ και να σας παρουσιάζουμε την αναφορά μας που αφορά εμάς και άλλα 900 άτομα που υπέγραψαν την αναφορά ε, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή σα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο προώθησης της συμμετοχής των Το άλλο είναι η υγεία και θέλουμε να επισημάνουμε μία από αυτές τις πτυχές, την υγεία και την προστασία της υγείας των πολιτών. Ολοκληρώνω ελπίζοντας ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι θεωρεί ότι είναι πιο σωστό για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι η διαδικασία επιπαραβάσει η κόψη της παραβίασης. Και δεύτερον, γιατί αυτό το έργο ε, είναι αντίθετο προς τους στόχους ε, της Οδηγίας 50 του 2008. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chairman. Um, well, here ε, this petition raises issues for... Κοιτάξτε, ε, τίθενται θέματα για τα οποία κατ' ουσίαν ε, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη και όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα, η περιβαλλοντική, η στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση έγινε τον Οκτώβριο του 2012. Η τροποποίηση ε, ελήφθη υπόψη και θα ληφθεί και περαιτέρω υπόψη ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές ε, δεν προέβησαν στην σχετική έκθεση ε, η... Ε, αφορά προγράμματα των διαδικασιών. Αλλά τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα και δεσμεύονται να εγκρίνουν προγράμματα μόνο ευτρέχει ε, μια διαδικασία επιπαραβάση στην περιοχή της Λομβαρδίας. Γνωρίζουμε ότι η ποιότητα του αέρα και της ατμόσφαιρας σε αυτή την περιοχή είναι πάρα πολύ κακή όπως ε, αναφέρθηκε ε, συνεχίζεται αυτή η διαδικασία και οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή των κρατών μελών και ως εκ τούτου ε, για μας πρόκειται για μία μεμονωμένη περίπτωση και για συστηματική αποτυχία σεβασμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Αυτή την τοποθέτηση σημαίνει ότι όσον αφορά στη συμμόρφωση ο σεβασμός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με το ότι δεν λαμβάνονται μέτρα αποζημίωσης και άμβλυνσης του προβλήματος, κυρίως για την κυκλοφορία. Μιλάμε για ένα σκι, όλα αυτά ε, δεν είναι λογικά και δεν ήθιστε, ε, δεν ε, συνηθίζεται ούτε καν να πηγαίνει κανείς σκι, όλα αυτά ε, δεν είναι λογικά και δεν ήθιστε. Ε, δεν συνηθίζεται ούτε καν να πηγαίνει πάρα πολλά τέτοια σχέδια τα οποία βρίσκονται στη φάση της ε, αδειοδότησης το Ασεγκράτε, το Αρογκά, Επιτροπή των Αφαρών. Η Ιταλία παραβιάζει νομοθεσία. Ο Υπουργό Γκαλέτη εκλήθη από τον Επίτροπο Βέλλα πριν από δύο περίπου εβδομάδων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, ήδη έχουμε θύματα γιατί η Ιταλία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό πρόωρων θανάτων. Η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή ε, και θέλω να παρακαλέσω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε την υγεία των ανθρώπων. Η Μάργαρετ. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Ελεονόρα. Δηλαδή, αν δει κανείς αυτή την ποιημένη ε, μελέτη επιπτώσεων, ε, όπως αναφέρθηκε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρέπει να συμφωνήσουμε, να δεχτούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, να υπάρχει ε, τουλάχιστον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά έχω και κάποια ανησυχία σχετικά με αυτή την οδηγία ε, ε, να υπάρχει τουλάχιστον η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά έχω και κάποια ανησυχία σχετικά με αυτή την οδηγία και ας ελπίσουμε ότι τελικά θα επικρατήσει και ο κοινός νους. Αυτό που λέει η Λεωνόρα φαντάζομαι ότι ο κοινό νους μπορεί τελικά να επικρατήσει και στην Ιταλία, στην εποχή μας τουλάχιστον. Όπως είπε η συνάδελφο και όπως γνωρίζετε είναι μία από τις ε, πιο ε, μολυσμένες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Έχουμε μεγάλη τύχη με τις Άλπεις από τουριστική σκοπιασμένα, αλλά αυτό μας δημιουργεί και ε, ένα ανώτατο όριο στη δυνατότητα ανακύκλωσης ε, του αέρα τη περιοχή και επομένως ο πολιτικό προσανατολισμός τη Ιταλία, τη Λομβαρδία και των ενδιαφερόμενων περιοχών όσον αφορά την πολιτική των υποδομών θα πρέπει να ε, ενδιαφέρεται και για την προστασία των συνθήκων που ήδη είναι επισφαλή ε, κυρίω για την ποιότητα του αέρα. Και βλέπετε ότι κυρίω ε, πλέον επενδύουμε σε έργα υποδομή, αυτοκινητοδρόμους, εμπορικά κέντρα και άλλα αντίστοιχα έργα τα οποία στο συνήθως και βλέπετε ότι κυρίω πλέον επενδύουμε σε έργα Αυτοκινητοδρόμου, αυτοκινητοδρόμου, εμπορικά κέντρα και άλλα αντίστοιχα έργα, τα οποία στο ε, συνήθως ε, είναι σε διαδικασία παραβάση για την παραβίαση και τις οδηγίες για την ποιότητα του αέρα και πρέπει να απαντήσουμε και στους πολίτες ε, που αμφισβητούν ε, τα θέματα αυτά διότι ε, στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν από αναπνευστικές ασθένειες ε, ή από στη χειρότερη από νεοπλασίας τα θέματα αυτά διότι στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν από αναπνευστικές ασθένειες ή από στη χειρότερη από νεοπλασίας καρκίνους που μπορεί φυσικά να αλλάξουν και την κοινωνική κατάσταση ενός ανθρώπου. Ε, είναι λοιπόν και κοινωνικό και κοινωνικο-οικονομικό το για την κυβέρνηση. Και ε, για τουριστικού λόγου, λοιπόν, όπω είπατε και εσεί, το είπε και η συνάδελφο, υπάρχει και μεταξύ των σχεδίων μία κότερα ε, ε, της αύξησης και τη μεγένθηκης. Δεν είναι το συγκεκριμένο έργο, αλλά και πολλά άλλα έχουν συζητηθεί για την περιοχή μου, τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε από κοινού και να τα επανακτολεί στην κυβέρνηση για να του πούμε ποιε είναι οι προοπτικέ που ε, ζητά η Ευρώπη για την περιοχή τη Λαμβαρδίας και ε, τα έργα υποδομή υποδομών. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ο για. Τέτοιου έργου. Αυτό είναι μια οικονομική απόφαση, αλλά υπάρχουν και θέματα που πρέπει να συναποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα είπαν οι προλαλήσαντε. Θα ήθελα να προσθέσω ένα στικτάρια 1500 στρέμματα καταστρέφεις μια καλώς λειτουργούσα οικογενειακή εκμετάλλευση γεωργική. Και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζουν οι τοπικές αρχές εκεί ότι, πώς να το πω, έτσι καλόβουλα ε, τους παρακολουθούμε και τους συνοδεύουμε και ε, προσέχουμε αν τηρούνται κάποιοι νόμοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το κάνει. Και ιδιαίτερα όταν καταλαμβάνεται ε, χώρο στη φύση, επιφάνειες, γες, αν είναι όλα σύνομα. Και εδώ υπάρχει και μια διχόνοια όταν τελειώσει το έργο. Καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω πώς ε, δρά. Βεβαίως ε, θα πρέπει να κινεί από την αρχή ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, δεν λέω ότι θα πρέπει να είσαι από χέρι καχύποπτος, αλλά όταν γίνεται τέτοιο έργο και υπάρχει και έχει κατασκευαστεί και εκ των υστέρων ερχόμαστε να διαπιστώσουμε ότι έχουν παραβιαστεί διάφορες νομοθεσίες, ε, το μόνο που διακυβεύεται είναι η καταβολή αποζημιώσεων χρηματικών. Από εκεί πέρα τίποτα. Βεβαίω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να πούμε στις αρμόδιες ιταλικές αρχές ξεκάθαρα ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς θα επαγρυπνούμε και θα φροντίσουμε να τηρούνται όλες οι διατάξεις. Τώρα, για την οικονομική σκοπιμότητα, εγώ τολμώ να την αφισβητήσω, πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί μου υπόθεση αυτό, αλλά ως ε, γεωργό, πραγματικά στεναχωριέμαι όταν φεύγουν οι γέε αυτές από τη Γεωργία. Και από την άλλη φτύνουμε αίμα στην Ευρώπη σε διάφορα ε, κράτη-μέλη ε, έχουμε την αντίστροφη κατάσταση ε, που καταστρέφουν δρόμους που έχουν κατασκευαστεί για να επανέλθει ε, στη φύση η γη αυτή. Ε, εντάξει, να κοιτάμε λοιπόν αν κτηρούνται πραγματικά οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες παντού. Ωραία. Και πάλι, από ό,τι φαίνεται, είμαστε όλοι σύμφωνοι πέρα από διαχωριστικές γραμμές πολιτικών ομάδων. με χαρά, από ό,τι φαίνεται, Είμαστε όλοι σύμφωνοι πέρα από διαχωριστικές γραμμές πολιτικών ομάδων. με χαρά προχωρήσουμε σε κάποια συμπεράσματα να ε, παρέμβουμε. Αυτή τη στιγμή ε, δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Προφανώς ε, και δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά στους ελέγχους. Η κατάσταση και το πρόγραμμα ως έχει τώρα προβλέπει έλεγχο και διορθωτικά μέτρα. Και νομίζω ότι τελικά αυτό μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Ως έχει τώρα προβλέπει έλεγχο και διορθωτικά μέτρα. Και νομίζω ότι τελικά αυτό μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Όσον αφορά ε, την κατάσταση όπως την παρουσιάσαμε σήμερα, σας είπα μπορούμε να παρέμβουμε. Πρόκειται προφανώς για ένα πρόγραμμα ε, που ε, δεν ε, είναι ότι θα φέρει ανάπτυξη στην Λομβαρδία. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προγράμματα στη Λομβαρδία και μάλιστα ε, δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου και από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το καθοριστικό στοιχείο. Να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη που να μην βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Μόνο να προσθέσω ότι αυτή η περιοχή τη δεκαετία του 60-70-80 ήταν καταστήματα. Αυτό δεν είναι σωστό κατά την άποψή μας. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας και την υγεία των παιδιών μας και γι' αυτό λοιπόν το θίξαμε. Yes, you are absolutely right. And this might... Έχετε το δίκιο. Μπορεί αυτό να είναι μόνη περίπτωση τώρα. Με αυτό το τελείως τρελό εμπορικό κέντρο και απίστευτο. Αλλά ε, το, πρόβλημα είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση στη ε, Λομβαρδία. Αυτή καθ' αυτή. Και έχουμε και πολλέ άλλε ε, αναφορά και θα στείλουμε επιστολέ στι αρμόδιες αρχές που ανάφερε η Ελεονόρα Εύη. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσουμε να μας ενημερώσει έως προς την ε, σημερινή κατάσταση και τα επόμενα βήματα. Στη... Ε, Έχουμε αναφορές για το ίδιο θέμα, τη 1253 και την 1353 για την ατμοσφαιρική ρήπαση στη Λομβαρδία. Και αφού κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά σε απότερο στάδιο, μπορούμε να τις εξετάσουμε από κοινού όλες τις αναφορές αυτές, το το οποίο έχει ξεφύγει λίγο από κάθε έλεγχο, όλα αυτά τα εμπορικά κέντρα, τα μολ. Εγώ δεν ξέρω γιατί ο κόσμος τα θέλει, εν πάση περιπτώσει και κατά πόσο χρειάζονται. Και όπως είπε και η Ελεονόρα, μπορεί να εστέφονται και κατά του τουρισμού. Στη Σουηδία και έχω συνηθίσει να κατεβαίνω πλαγιέ ε, στον καθαρό αέρα, με τον ήλιο. Αλλιώ ψευτοσκή είναι αυτό είναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, επιστρέψτε στην όμορφη αυτή γωνιά της Ευρώπης που είναι η πατρίδα σας και ελπίζουμε κάποιες περιοχές να παραμείνουν προστατευμένες. Πάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά, η παριθμό 27. Αποουσιάζει ο αναφέρον, ε, πλην όμως παρευρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σφάρκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Η αναφορά αφορά την προσφυγή του κυρίου Χατζησάβα ε, για άδικη διέμβη σε θέματα εθνικής δικαιοδοσίας. Είδαμε λιγάκι και το θέμα του υπενιγμού από ε, πληροφορίες για το ε, τι είδους ε, πρόγραμμα ήταν αυτό. Δεν αναφέρεται στην χρήση σε τίποτα. Και για το λόγο αυτό ε, δεν μπορούμε κι εμείς να βρούμε δικογραφία, όλα τα σχετικά έγγραφα και κατέληξε και η Όλαφ ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στο ότι και η ίδια πρέπει να επιληφθεί του θέματος να διεξάγει έρευνα. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν τουλάχιστον. Ο Πίτα. Ε, θα του εξηγήσουμε γιατί ε, κλείνει αυτή η αναφορά. Αν ο αναφέρον είχε συγκεκριμένα στοιχεία θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε ανοιχτή. Αλλά πολύ σωστά είπατε στην πρώτη σας παρατήρηση ότι δεν μπορεί κανείς να παρεμβαίνει σε εσωτερικά θέματα δικαιοσύνης και δεύτερον ε, ο αναφέρον θα ενημερωθεί αν δεν συμφωνεί μπορεί να... μπορούμε να πούμε ότι κλείνει αυτή η αναφορά. Αυτή είναι μια αναφορά του 2013. Ε, τότε εγώ δεν ήμουνα πρόεδρος ε, και νομίζω ότι με μονομένη περίπτωση και επειδή ε, πρόκειται για κατάχρηση ενωσιακών πόρων παραπέμφθηκε στην Όλαφ και δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να κάνουμε οτιδήποτε με αυτή την αναφορά. Ας την κλείσουμε λοιπόν. Πολύ ωραία. Και πάμε στο επόμενο θέμα που είναι του αναφέροντα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πράσις. Και για μένα είναι τιμή. Ο πρόεδρος Μακρόν προτείνει διαβουλεύσεις με τους πολίτες, για τους πολίτες και θα πρέπει ε, ε, να γίνει αποκεντρωμένη συζήτηση ε, δημοτικούς συμβούλους και το καταθέτει η Ένωση Ευρωπαϊστών και Φεντεραλιστών της Ισπανίας. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Τι λέμε, να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δίκτυο εκεί ολοκλήρωση και ιστορία της, αξίες, πολιτικές και δικαιώματα της Ένωσης ε, προκλήσεις ε, κλπ. Τον Ευρωπαίο πολίτη, όπως έλεγε και ο δικός χάρτης Βρατισλάβα, το Σεπτέμβριο του 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απαντάει ότι υπάρχουν οι έδρες Ζαμονέ, βεβαίως είναι πολιτικού, στα χωριά, όπως πολύ ωραία λέει το σημείο 9 της ε, ε, ανακήρυξης ε, της Συνόδου Κορυφής των χωρών του Νότου, 10 Ιανουαρίου. Η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λέει τίποτα ως προς τη δυνατότητα να διερευνήσουμε με πολύ λίγα λεφτά ε, το δυναμικό που έχουν χιλιάδες δημικοί κοινότητες στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη του 2017 και στην παράγραφο 28 λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει με στόχο την ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη μέχρι να ε, δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό το Κοινοβούλιο με την επιφύλαξη των προηγουμένων ε, να... Η... όχι. Συγγνώμη, πρώτα πρέπει να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα κι εγώ. Ο κύριος Αγγελιανός, παρακαλώ. Yes, thank you. Um... Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα και να επισημάνω ότι συμφωνούμε απολύτως και ε, συμφωνούμε με την άποψη ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτό το σκοπό. Ε, πιο συγκεκριμένα το βραβείο Αλτιένο, Αλτιέρο Σπινέλη, το οποίο δόθηκε για πρώτη φορά το 2000 και μάλιστα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δόθηκε μάλλον για πρώτη φορά το 2017 που εδώ και αρκετά χρόνια ε, στόχο έχει να ε, προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες ε, και να βελτιώσει ε, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη ε, διαδικασία ε, χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις από τότε που παρουσιάστηκε αναφορά, τους τελευταίους μήνες δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτές είναι πρώτον ότι το φθινόπωρο 2017 η Ευρωπαϊκή Επιστόχο μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αποτελέσματα, προσφέρει ε, ενίσχυση και προστατεύει και αυτή ε, η εκστρατεία ενημέρωσης και ε, επικοινωνίας ξεκίνησε το φθινόπωρο. Άσμους πλάς, Έχω φέρει και ένα αντίγραφο εδώ για να λάβει υπόψη του ακριβώς αυτή τη διάσταση που προτείνετε κι εσείς. Μονέ, μέσω της επικαιροποιημένης ε, εκδοχής ε, που έχουμε τις διάφορες δραστηριότητες Ζαμονέ, τις λεγόμενες έδρες Ζαμονέ, τα δίκτυα αριστείας Ζαμονέ, ε, προγράμματα Ζαμονέ, στήριξη προς για δημάρχους ε, και συμμετοχή ε, δημάρχων και ε, δημοτικών συμβούλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα βρείτε λοιπόν ότι υπάρχει πλέον τέτοια διατύπωση για τις απαιτήσεις για τους δικαιούχους των δραστηριοτήτων Ζαν Μονέ, τους δικαιούχους των διαφόρων δραστηριοτήτων Ζαν Μονέ να να συνεργαστούν με πολίτες και την κοινωνία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο και να υπάρχει και καθηγητές δηλαδή των, ε, που θα κατέχουν την έδρα Ζαμονέ, ε, θα πρέπει να ε, οργανώνουν δραστηριότητες, διαλέξεις, εργαστήρια κλπ. με διδάσκοντες σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή με δημάρχους και δημοτικούς στασί, αυτή την προσέγγιση και την ενημέρωση των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών και σε επίπεδο ε, υποχρεωτικής ε, παιδείας ε, στα μελλοντικά προγράμματα. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι αν επενδύσουμε για καλύτερη παιδεία, καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη ε, έμπνευση προς τους πολίτες ε, για αυτό το οποίο αποκαλούμε Ευρώπη, θα πρέπει να ξεκινά ε, από την πρώτη σχολική ηλικία και εξετάζοντας τι να κάνουμε για τα μελλοντικά προγράμματα, το εφαλτήριό μας είναι ότι αυτή η διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα η διδασκαλία, η ενημέρωση για την Ευρώπη σε επίπεδο υποχρεωτικής ε, ε, παιδείας ε, ήδη από την πρώτη υποχρεωτικής στα μελλοντικά προγράμματα. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι αν επενδύσουμε για καλύτερη παιδεία, καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη ε, έμπνευση προς τους πολίτες ε, για αυτό το οποίο αποκαλούμε Ευρώπη, θα πρέπει να ξεκινά ε, από την πρώτη σχολική ηλικία και εξετάζοντας τι να κάνουμε για τα μελλοντικά προγράμματα, το εφαλτήριό μας είναι ότι αυτή η διάσταση θα πρέπει να ενισχυθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα η διδασκαλία, η ενημέρωση για την Ευρώπη σε επίπεδο υποχρεωτικής ε, ε, παιδείας ε, ήδη από την πρώτη σχολική ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πλήρη ε, παρουσίαση και για το προσωπικό πάθος που επιδείξατε. Έτσι πρέπει να είναι από τα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντως, λέει η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Και κατηγορηματικά τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί όπως είπε και η Πρόεδρος, ήταν πάρα πολύ πλούσια αυτά που μας είπε με καινούργια στοιχεία, αλλά και κατά την άποψή μου φαίνεται ότι υπάρχει προσωπική δέσμευση και πολύ καλή εστίαση. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι εξακολουθεί. Γίνεται ρητή αναφορά στην εντολή μας. Όπως αναφέρθηκε και η πρόσφατη έκθεση για την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, που είναι έκθεση επί της Ευρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητούμε ρητά ε, να είναι δραστηριοτήτων, να συμμετέχουν οι ίδιοι οι πολίτες στο Δήμο τους για να τους δώσουν έτσι μια νέα πνοή και ένα περιεχόμενο στις δραστηριότητες αυτές. Δηλαδή ε, δεν θα πρέπει να είναι παθητικοί αποδέκτε κάποιων μηνυμάτων οι πολίτες, να συμμετέχουν και να ενεργούν και οι ίδιοι. Ε, πολύ καλό αυτό που μας είπατε για την ε, ενημέρωση και επικοινωνία στους ε, δύο επιτρόπους που ασχολούνται με θέματα ηθαγένειας και ιδιότητας του πολίτη, την κυρία Γιούροβα και στον κύριο Αβραμόπουλο δηλαδή, λέγοντας ότι υπάρχει έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει εγκρίνει κάποια πράγματα. Και επίσης η Επιτροπή Πολιτισμού γνωμοδότησε στη δική μας έκθεση και ξεκαθάρισε μετα... τι κάνουμε και πώς συνεργαζόμαστε εμείς από την πλευρά μας. Και όταν θα έχουμε μια πιο φρέσκια ε, απάντηση για το τι θα γίνει στο μέλλον, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να δούμε πώς μπορεί ο πολίτης από αυτό το ανοιχτό παράθυρο που είναι η Επιτροπή Αναφορών να προχωρεί συμμετοχή και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Thank you very much. And now I will try something. Very often, very... Πολύ συχνά είναι αδύνατο οι συνάδελφοι να προφέρουν το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Μπεθέρα και θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να πω και εγώ ότι και εμείς θα θέλαμε να παραμείνει αυτή η αναφορά και ευχαριστούμε βεβαίως τον Ταμιάν Μαθίας για την πρότασή του και για την εξαιρετική εξήγηση που μας έδωσε. Μέσω της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Δήμου, στην οποία στον οποίο αναφερθήκαμε πάρα πολλές φορές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπιστώνουμε ότι έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες αυτού του όμορφου οικοδομήματος ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε πάρα πολλά μέτρα στα τομέα της επέκτασης και της σημασίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ιδιαίτερα σε τοπικό και σχολικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ευρύτερους πολιτιστικούς χώρους, για παράδειγμα, ε, μέσω του αθλητισμού, στον οποίο, ε, μέσω του οποίου η Ευρώπη θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτό τον κοινό δήμο, σε αυτή την κοινή ε, συμμετοχή και άμυλα πολλές φορές διάφορα κινήματα δημιουργήθηκαν χάρη σε μεγάλα έπι, ακόμα και στον αθλητισμό. Η Ισπανία, για παράδειγμα, δεν συμμετέχει κάπου αλλού πέραν από το μάλλον συμμετέχει σε όλα εκτός από τον γκολφ. Ε, εγώ θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη θέση στο σχολική εκπαίδευση ε, και εγώ ε, έκανα κάποιες σπουδές σε ευρωπαϊκά σχολεία και σε κάποια σχετικά γνωστά σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα ε, θα πρέπει η πρόταση να ε, αναλάβουν οι δήμοι, δηλαδή οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι ε, όλη τη Ευρώπη κάποια πράγματα να προωθήσουν, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ιδέα. Και νομίζω ότι συνάδει και με την